Δουλεύει λοιπόν το σύστημα. Διαρωτάται ο πρόεδρος. Σας καλωσορίζω. Είπα χτες λόγω του blackout το θέμα το οποίο ασχοληθήκαμε ε, αναβλήθηκε και γι' αυτό προσπαθούμε σε συνεργασία με την γραμματεία να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Ίσως ε, να επανέλθουμε στα θέματα που μας απασχολούν την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα σας ενημερώσουμε. <coughs> Ε, λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τώρα να εκμεταλλευτούμε την ώρα που έχουμε μπροστά μας. με το Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο καλωσορίζουμε having here... με τον Υπουργό Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι τιμή μας που είναι παρόν εδώ σήμερα υπεύθυνο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Έρικ Χόλτερ, ο οποίος συνοδεύεται από τον πρέσβη Κενάρντ και από τα μέλη της συνοδείας τους. Όλους τους καλωσορίζουμε λοιπόν στις Βρυξέλλες στοχεύουμε να ακούσουμε από τον κύριο Γενικό Εισαγγελέα ή Υπουργό Δικαιοσύνης την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο διάλογος και η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε στα δικαστικά θέματα. Είναι πολύ σημαντικός ο, τομέας αυτός σε αυτή τη φάση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας η οποία εμπλέκεται σε πάρα πολλά θέματα όπως τις διαπραγματεύσεις για τα PNR και για τη Γενική Συμφωνία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Είναι παρόλα αυτά μια ευκαιρία για όλους εμάς να δούμε σε ποια φάση βρίσκονται οι συμφωνίες τις οποίες διαπραγματευθήκαμε επί μακρόν και τις οποίες υιοθετήσαμε το 2003 και επικυρώθηκαν το 2009 και τέθηκαν σε λειτουργία το 2010 και στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρώπη για την αμοιβαία νομική σύνδρομη και τις διαδικασίες έκδοσης. Θα υπάρξει λοιπόν δυνατότητα για να συζητήσουμε τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο σημαντικές συμφωνίες και για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών για τις α, τραπεζικές συναλλαγές και για την αμοιβαία νομική συνδρομή. Αρρωγή. Αρρωγή και για τον τομέα επίσης όπως προείπα τον, της έκδοσης. Ε, εν πάση περιπτώσει ελπίζω την επόμενη ώρα να ακούσουμε από τον κύριο Έρικ Holder για τα επόμενα 10 ή 15 λεπτά και μετά θα ξεκινήσει ένας πρώτος γύρος ε, ανταλλαγών ε, με τους συντονιστές που θα πάρουν το λόγο πρώτοι για δύο λεπτά και θα υπάρξει χώρος ε, να απαντήσει, χρόνος να απαντήσει ο Γενικός εισαγγελέα και μετά ε, θα ακούσουμε για ένα λεπτό τις παρεμβάσεις των μεμονωμένων μελών που έχουν συγκεκριμένα θέματα ίσως να θέσουν γύρω από τα υποσυζήτηση προβλήματα. Εσείς που θέλετε να πάρετε το λόγο ενημερώστε μας για να γνωρίζουμε ποιοι είστε. Και θα υπάρξει λοιπόν όπως είπα ένας πρώτος γύρος δύο λεπτά για τους συντονιστές και ένα λεπτό για τον μεμονωμένο απλό βουλευτή μετά. Αυτός θα είναι ο μοναδικός τρόπος ε, για να προχωρήσουμε λόγω ακριβώς της έλλειψης χρόνου η οποία χαρακτηρίζει τον ε, κύριο Υπουργό. Έχετε το λόγο Καλή σας μέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Τιμή μου είναι να προσφωνήσω τα αξιότιμα εξωχαμέλη αυτής της Επιτροπής ε, και να μιλήσουμε για τα θέματα των ευθυνών, τα θέματα των ευθυνών που συμμεριζόμαστε. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργός Δικαιοσύνης είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας με πολλούς από εσάς και με ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο καθώς επίσης και με Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών από πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση των ΗΠΑ των σχέσεών μας που επιθυμούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μου. Από τότε που ανέλαβα το αξίωμά μου, καλλιέργησε αυτές τις σχέσεις όσον αφορά τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και κάθε έξι μήνες είχαμε τέτοιου είδους επαφές και κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας θα έχουμε τέτοιου είδους συναντήσεις. Είναι προνόμιο να είμαι μέρος αυτής της συνεργασίας και να βλέπω τις ειδικέ σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των εθνών μας επί τόσα έτη, που βοήθησαν να προστατεύεται η συλλογική ασφαλειά μας, η ευημερία μας, καθώς επίσης και οι πολιτικές ελευθερίες μας. Και όπως κάθε ένας από εσά, έτσι και εγώ θέλω να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια με αυτές τις επιδόσεις. Και αυτό με φέρνει εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες και ενώπιόν σας. Και εξ ονόματος του Πρόεδρου Ομπάμα και του Αμερικανικού λαού θέλω να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε να προσέλθω σε εσά και που με καλωσορίσατε σε αυτή την όμορφη πόλη. Και ελπίζω και ευελπιστώ πράγματι ότι έχω εμπιστοσύνη ότι όπως και τόσες φορές αυτό, αυτή η συνάντησή μας θα δώσει καρπούς όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την συνεργασία και τονίζω με αυτή την κοινή συνεργασία υπέρ κοινών σκοπών και με καλές προθέσεις ε, και με αμοιβαίο σεβασμό και πάντα με αμοιβαία συνεργασία είμαστε επιτυχείς στην οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς κόσμου. Ταυτοποιήσαμε, εντοπίσαμε και αποδιαρθρώσαμε διεθνή δίκτυα του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, ε, εμπορίας ανθρώπων ε, και πολλές, πολλά τέτοια προγράμματά τους και προσπάθειές τους. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάθε έκφραση βίας, κυβερνοέγκλημα, ε, περίπτωση ε, διαφθοράς όσον αφορά κυβερνητικούς εκπροσώπους και εκμετάλλευση παιδιών. Και ενώνοντας ε, τις προσπάθειές μας πάντα είμαστε υπέρ των πολιτικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και καταφέραμε να προστατεύσουμε σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα. Στην καταπολέμηση του εγκλήματος και του, της διαφθοράς πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύουμε την ιδιωτική σφαίρα, την ιδιωτική ζωή των πολιτών μας. Υπάρχουν τρεις ε, συμφωνίες που πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Η ε, ΕΠΑ Ευρωπόλ, ΕΠΑ Eurojust και η ε, συμφωνία για την έκδοση και παράδοση όσον αφορά τις ε, περιπτώσεις εγκλημάτων μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι τρεις συμφωνίες έχουν δώσει την ευκαιρία σε πολλές ανταλλαγές πληροφοριών και πολλές κοινέ δράσεις και πολλές ε, εξεταστικές ε, δράσεις και ανακρίσεις που έδωσαν την ευκαιρία να προστατευτούν πολίτες και να προστατευτεί και η ιδιωτική του ζωή. Νομίζω ότι είναι υποδείγματα, λαμπρά υποδείγματα επιτυχίας σε σχέση με την κοινή μας συνεργασία. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια πρόταση ότι υπήρξε κάποτε, υπήρξε ποτέ μια οποιαδήποτε παραβίαση, έστω και ατομική παραβίαση δικαιωμάτων μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να βασιζόμαστε πάντα στα πραγματικά γεγονότα και όχι σε υποθετικά γεγονότα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα γιατί καταφέραμε να πετύχουμε ε, συνεργαζόμενοι με την Eurojust και την ε, Europol και τους ε, εκπροσώπους των αστυνομικών δυνάμεων όσον αφορά ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα καταφέραμε να κλείσουμε ένα μεγάλο δίκτυο παιδικής πορνογραφίας και εκμετάλλευσης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών παιδιών. Αυτό το οποίο θα ήταν μια ατομική σύλληψη οδήγησε σε μια συλλογική και ε, ανάληψη δράσης κατά 20 κατηγορουμένων σε διάφορες χώρες. Καταφέραμε να σώσουμε παν, περίπου 50 παιδιά, 50 παιδιά, τα πιο ευάλωτα από, όλα, από όλους τους πολίτες, εκτεθειμένα σε αυτά τα εγκλήματα. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα από τις θετικές επιπτώσεις της κοινή προσπάθειάς μας και δράσης μας όσον αφορά τις, ε, ε, τα δικαιώματα δικαιώματα και της ελευθερίας. Τίποτα δεν είναι τόσο κατεπήγον όσο η καταπολέμηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Και ακριβώς αυτό μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαμε την δέκατη επέτειο της πιο τρομακτικής ε, απόπειρας τρομοκρατίας ε, του 2001 ε, που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 της, ε, στην, την 11η Σεπτεμβρίου και όπου είχαμε τόσα θέματα που χωρίς κανένα νόημα δολοφονήθηκαν. Είχαμε δεκάδες Ευρωπαίους, ε, Γάλλους, Γερμανούς, Ιρλανδούς, Ιταλούς, ε, Λιθουανούς, Ολλανδούς, Πορτογάλους, Πολωνούς, Ρουμάνους, Ισπανούς, Σουηδούς, Βρετανούς, καθώς και Βέλγους που ήταν θύματα αυτής της τρομοκρατικής, ε, αυτού του τρομοκρατικού πλήγματος. Ε, συνήρθαμε ενωμένη σε αυτή την επέτειο με την κοινή θλίψη και πένθος αλλά και την κοινή απόφαση και σθένος να συνεργαστούμε ως εταίροι, ως σύμμαχοι, να αντιμετωπίσουμε τις απειλές που έχουμε ενώπιόν μας σε μια ιστορική συγκυρία ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τις κοινέ αρχές και αξίες μας. Και σαν άμεση αντίδραση στην 11η ε, ε, Σεπτεμβρίου συνήθαμε και έχουμε αυτό το πλαίσιο των συμφωνιών και έκδοσης ε, για να καταδείξουμε στον κόσμο ότι αυτή η εταιρική σχέση υπέρ τη ε, ελευθερίας και των ελευθεριών των πολιτών μας και υπέρ του σθένου μας ε, να είμαστε ενωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, τα τελευταία χρόνια θυμηθήκαμε και στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη και στην Καμπάλα και στην Βομβάη με τα τρομοκρατικά πλήγματα και στην Αμπούζα πιο πρόσφατο πλήγμα ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε πραγματικά πραγματικές ε, και χειροπιαστές ε, απαιτούν την διαρκή προσοχή μας, εγρήγορση διαρκή και συνεργασία μας. Έχουμε ενώπιόν μας λοιπόν μια ευκαιρία. Ευκαιρία να σημειώσουμε πρόοδο περαιτέρω συνεργαζόμενοι στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας αλλά υπερασπιζόμενοι τις πολιτικές ελευθερίες επιπλέον και υπερασπιζόμενοι και την προσωπική ζωή των πολιτών μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά και επεκτείνοντας τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά της ΕΠΑ και την ε, Ευρωπόλ, την ΕΠΑ, την Eurojust μέσω αυτών των συμφωνιών στο πλήρες εύρο των διατάξεων και κανονισμών όσον αφορά τα, τη δράση μας ε, μεταξύ ε, ΕΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Αναφέρθηκα στις ευρύτερες διασφαλίσεις ε, που δίνονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεν γνωρίζω να υπάρχουν οποιασδήποτε παραβιάσεις αυτών των εγγυήσεων. Έχουμε μια ευκαιρία λοιπόν να παγιώσουμε, να θεμελιώσουμε αυτές τις εγγυήσεις σε τέτοιες συμφωνίες για την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων που θα συνεισφέρουν υπέρ τη ευημερίας των πολιτών μας. Είναι ένα φιλόδοξο και πολύ ε, θα έλεγα ε, μεγαλόπνο εγχείρημα διότι πέρα από τι επιμέρου ανταλλαγέ ε, στοιχείων για την καταπολέμηση τρομοκρατία, όπως αυτά που αφορούν τα στοιχεία των επιβατών αεροπορικών εταιριών και των προγραμμάτων που έχουμε υποεξέλιξη έχουμε κάθε λόγο να ευελπιστούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα ευδοκιμήσει λαμβάνοντα υπόψη ότι οι διατάξει που έχουμε διαπραγματευτεί σε σχέση με τι συμφωνίε αυτέ θα πρέπει να είναι αποτελεσματικέ, προστατεύοντα την προσωπική ζωή μέσα στα συστήματα δικαίου και τη ένωμη τάξης. Ενώ δεν μπορώ να επιστρέψω σε λεπτομέρειε όσον αφορά τι τρέχουσε διαπραγματεύσει, μπορώ να σας πω ότι οι διαπραγματευτές μας, αμφωτέρωθεν του Ατλαντικού, συνεργάζονται από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις τον Μάρτιο, συνήθαν και είχαν και βιντεοδιασκέψεις εννέα φορέ. Δεκάδες ωρών ανάλωσαν και επένδυσαν σε αυτά τα θέματα, στην εξέταση θεμάτων που βρίσκονται λίγο πριν από την ολοκλήρωση ε, και την ευδοκίμηση. Και για την, ε, το πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια από τα θέματα που αποτελούν θέματα κλειδιά της προσπάθειας αυτής. Πρώτα απ' Ενώ είναι σωστό να έχουμε ε, και να τονίζουμε αυτέ τι κοινέ αξίε και αρχέ για τα νομικά μα συστήματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι βασικέ νομικέ διαθρώσει και δομέ και οι διαφορετικοί κανονισμοί και διατάξει όσον αφορά τι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν κάποιε διαχωριστικέ γραμμέ. Δεν είναι δυνατόν να συγχωνευτούν ή να επιβληθούν διατάξει από το ένα νομικό σύστημα στο άλλο. Αντίθετα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάθε ένα από τα δικά μα ξεχωριστά συστήματα προστατεύουν τι πολιτικές ελευθερίες και την ιδιωτική ζωή και σφαίρα, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Αυτή είναι η αμοιβαία αναγνώριση που πρέπει να αποτελεί την βάση, τα θεμέλια για να προχωρήσουν αυτές οι συμφωνίες. Αντί να έχουμε μια προσέγγιση σημείο ανά σημείο, θα πρέπει να πούμε σε σχέση με την γενική μας προσέγγιση ότι θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές οι διαδικασίες οι οποίες θα συμφωνηθούν και ε, λειτουργούν ήδη. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι οι διαφορετικές ε, ιστορίες ε, και τα διαφορετικά προηγούμενα μπορούν να οδηγούν σε διαφορετικά νομικά πλαίσια. Προστατεύοντας όμως πάντα τις ίδιες αρχές και αξίες όσον αφορά τους ανθρώπους στις οποίες πιστεύουμε. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τις διαφορές του δικαίου και της νομοθεσίας και νομολογίας όσον αφορά τη ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε ότι τα κράτη-μέλη και η ΕΕ κατάφεραν να ανταλλάξουν και να προστατέψουν στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα μέσα σε αυτήν την προσπάθεια υπέρ της ασφάλειας. Θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να τονίσουμε αυτές τις κοινές, αυτά τα κοινά πεδία και κοινά θεμέλια όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Όχι μόνο για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και για τη διασφάλιση διαφάνειας στις δράσεις μας. Παράδειγμα, στη ΗΠΑ. Ε, ο νόμος για την ελευθερία για τα θέματα πληροφόρησης δίνει την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση ε, σε τέτοια στοιχεία οι πολίτες άσχετα από την προέλευση ή την υπηκότητά τους και φυσικά η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αρνούνται την ε, ατομική πρόσβαση σε κάποια στοιχεία αν αυτά είναι διαβαθμισμένα και είναι αναγκαίο να τηρούνται μυστικά όπως για παράδειγμα για κάποιες ε, διοκτικές, ε, την ανάληψη διοκτικών δράσεων. Θα πρέπει λοιπόν χωρίς να θυσιάζεται η δημόσια ασφάλεια να ε, σεβόμαστε αυτές τις αρχές. Δεν έχω υπόψη να υπάρχει κάποια άλλη χώρα που να έχει τόσο ισχυρό πλαίσιο όσο αυτό το νομικό πλαίσιο που έχουν οι ΗΠΑ για την ελευθερία, το νόμο για την ελευθερία της όσον αφορά την πληροφόρηση. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και την καταδίωξη των σημαντικών περιπτώσεων εγκλήματο, οπουδήποτε και αν αυτά έχουν λάβει χώρα λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την αμοιβαία νομική αρρωγή, την αμοιβαία νομική συνδρομή, προστατεύοντας πάντα, αναλαμβάνοντας τέτοια δράση τα δικαιώματα των πολιτών μας. Και αυτό επειδή υπάρχουν αυστηρότατες, αυστηρότατοι περιορισμοί όσον αφορά τη ΣΥΠΑ αλλά και την Ευρώπη για την διασφάλιση αυτών των προσωπικών δεδομένων των πολιτών μας. Αυτή η δέσμευση υπέρ της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, αμφωτέρωθεν του, των όφεων του Ατλαντικού, δίνει μια καθοριστική αρχή που είναι καταλύτης ε, και που είναι ξεχωριστή μεταξύ όλων των ε, κοινών αρχών και αξιών που μας ενώνουν. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αξίες για τον ίδιο τον πρόεδρο Ομπάμα, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και για μένα τον ίδιο προσωπικά ως Υπουργό Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να προσέλθω σε εσά και να σας προσφωνήσω εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των, ε, του λαού μας και ε, δίνοντας συνέχεια σε αυτή τη δέσμευση υπέρ των δικαιωμάτων, υπέρ όλων η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιδιαίτερες ε, ελευθερίες που αναγνωρίζουμε και η ιδιαίτερη αξία που δίνουμε σε, αυτή, σε αυτές τις ελευθερίες, πολιτικές ελευθερίες των πολιτών μας. Η θα είναι πάντα στο στο πλευρό σας ως σύμμαχος, ως εταίρος με τα σημερινά συστήματα τα οποία πρέπει να αντανακλούν την ανάγκη να προστατέψουμε τους πολίτες, αλλά υπόψη και το ίδιο το Σύνταγμα που θεσπίζει ένα, μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση με συγκεκριμένες ε, εξουσίες και πάντα μέσα σε ένα σύστημα ελέγχου των εξουσιών αυτών. Και με αυτόν τον τρόπο βλέποντας ε, ότι με αυτόν τον τρόπο ε, συνεχίζουμε τη δράση μας και μέσω της δικαιοσύνης και η διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα, μια συνταγματική επιταγή. Για πάνω από δύο αιώνες οι Αμερικανοί ε, προσπαθούν και δίνουν μάχη για την ε, υπεράσπιση αυτών των αξιών. Είναι ε, ακριβώς ο σωστός προσανατολισμός για το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα στι ΗΠΑ. Συζητώντας αυτά τα θέματα όχι μόνο οι πολίτες των ΗΠΑ κατανοούν τις ανησυχίες και τα μελήματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι τα πράγματα αυτά ε, δεν, αναμένουν, δεν παραμένουν χωρίς να αντανακλούν ε, και την ίδια την ε, νομική τάξη. Οπότε πρέπει να δούμε την αντιστοιχία των αρχών με τις δράσεις. Και θα πρέπει εδώ η αποκάλυψη περιπτώσεων παραβίασης ή παράβασης εξουσίας ή δικαίου να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί. Και πιστεύω ότι <clears throat> σε καμιά άλλη χώρα και σε σχέση με το 2009 και 2010 που είχαμε ε, ε, προσάξει τη δικαιοσύνη κατηγορούμενους ε, που ουσιαστικά είχαν ακριβώς παραβεί αυτές τις αρχές, δηλαδή την χωρίς ε, οποιαδήποτε ε, λόγο πρόσβαση σε ε, στοιχεία και παραβίαση των αρχών της προστασίας ιδιωτικής ζωής. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά λαμβάνουμε εμείς υπόψη τα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Και έτσι η ένταξη αυτών των στοιχείων μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας συλλογής στοιχείων και δεδομένων δεν έχει προηγούμενο στον κόσμο. Και διασφαλίζοντας ένα υψηλότατο επίπεδο <clears throat> ώστε σε σχέση και με το Κογκρέσο όσον αφορά τις ε, έρευνες ε, και την ανάληψη δράσης για να υλοποιείται από την κυβέρνηση αυτή η σημαντικότατη ευθύνη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ε, αντίθετα σε ό,τι πιστεύουν πολλοί οι κανόνες και κανονισμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη ΣΥΠΑ έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο όσον αφορά για παράδειγμα τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ε, και έχουμε τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις ε, για να διεξάγονται τέτοιες έρευνες. Επίσης, ε, κανόνες και κανονισμοί όσον αφορά την λογοδοσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους πληροφορίες, παράδειγμα τεστ DNA και ε, ανάληψη σχετικής δράσης, ε, καθώς επίσης και προστασία ε, για όλους τους πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, δεν εκπλήσει κανένα ότι οι επαΐοντες και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από πολιετή εξέταση και συζήτηση αυτών των θεμάτων, κατέληξαν στο ότι παράθεμα έχουν κοινό στόχο στην κοινή αυτή δέσμευση για την προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ε, σφαίρας, της ιδιωτικής ζωής κατά τη συλλογή δεδομένων. Τέλος παραθέματος. Έτσι πρέπει να είναι υποφελείς οι συμφωνίες μας ανταλλαγής δεδομένων και στοιχείων όπως είπα Europol, είπα Eurojust ε, και ε, των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων ταξιδιωτών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα ενώ συνεχίζονται αυτές οι διαπραγματεύσεις ευελπιστώ ότι από αυτή τη συνεργασία θα έχουμε ένα κοινό ισχυρό ισχυρό δεσμό που θα αναγνωρίζει ότι τα συστήματα τα οποία έχουμε πρέπει να προστατεύουν αποτελεσματικά αυτά τα δικαιώματα παρότι είναι διαφορετικά τα συστήματά μας και έτσι θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα μέγιστα ωφέλη από μια γενική συμφωνία που θα θέτει μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυτές τις αρχές. Είναι μια πρόκληση. Άσχετα ποια είναι η πρόκληση και ποιες είναι οι διαφορές όσον αφορά την χρονική συγκυρία και τις παρεκκλήσεις, πάντα θα είμαστε ενωμένοι και εταίροι. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και εταίροι. Μα ενώνουν οι αρχέ και οι αξίε μα. Οι κοινέ ευθύνε, η υπευθυνότητα που έχουμε να προστατεύσουμε τι πολιτικέ ελευθερίε και τα δικαιώματα των πολιτών μα. Και να συνεχίσουμε μέσα σε μια δυσχερέστατη συγκυρία παγκόσμια να συνεχίσουμε την κοινή μα πορεία. Αυτή είναι η πρόκληση. Και θέλω να σα ευχαριστήσω και όχι μόνο να κάνουμε αυτό το οποίο είναι αναγκαίο, αλλά αυτό το οποίο είναι σωστό και δίκαιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Τώρα θα προσέξω τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κι εμείς. Ε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την... τα ενθαρρυντικά σας λόγια όπως τονίσατε μοιραζόμαστε κοινέ αξίε, την δέσμευσή μα να αποκαταστήσουμε και να διατηρήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στι ανάγκε τη δικαιοσύνη και στι ανάγκε προστασία τη προσωπική σφαίρα των πολιτών μα. Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί και ακόμα πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή μας των Θεμελιωδών Ελευθεριών και θα εξετάσουμε, θα εγγύψουμε και στις ε, λεπτομερείς πτυχές των ε, συμφωνιών που έχουμε υπογράψει και που διαπραγματευόμαστε. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ομάδα ειδικών καθηκαοντών, μια task force από το 2009 για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών ε, δικαστικής αρρωγής και εκδόσεως. Έχουμε κοινέ ομάδες τώρα, έχουμε και ε, ανταλλαγή πληροφοριών και τόσες άλλες πτυχές οι οποίες θα, έχουμε τη δυνατότητα, θα έχουν τη δυνατότητα μάλλον να συζητηθούν στις πρώτες συνεδριάσεις. Όπως είπα τώρα, δύο λεπτά ο κάθε συντονιστής από κάθε πολιτική ομάδα και μετά θα προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ρωτήσεων που ε, θα διαθέσω ένα λεπτό στο κάθε, στον κάθε βουλευτή. Και σας παρακαλώ να τηρήσετε τα χρονικά αυτά όρια, διότι οι ανηλυμένες υποχρεώσεις του ε, κύριου Υπουργού είναι βέβαια πάρα πολύ ε, ε, Ο κύριος Βέμπερ συντονιστής του Λαϊκού κόμματο. Κύριε Υπουργέ, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, περιμένω ε, λίγο για να φορέσετε τα ακουστικά σας. Αυτό είδα και εγώ. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Θα δώσω εγώ τα ακουστικά μου στον ε, κύριο Υπουργό. That's a cooperation translator, yes. Okay. Καλώς ήρθατε, σας ευχόμαστε εγκάβιο, καλώς ορίσατε στον Υπουργό Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ήθελα πρώτα να τονίσω ότι σε όλη την Ευρώπη ξαναστοχαστήκαμε τα φρικτά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 2001, προ μιας δεκαετίας, που ήταν για, απαιτέλεσαν βαθιά τομή και στον τρόπο ζωή μα και τον δικό σα και τον δικό μα. Εξ ονόματο τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο θα σα ευχαριστήσω για την δεκαετή συνεργασία και στην, στον αγώνα κατά τη τρομοκρατία που ωφέλησε και τι ευρωπαϊκέ χώρε. Έχουμε τώρα ορισμένα θέματα επιτάπιος τα οποία μας συγκινούν. Το πιο σημαντικό είναι το θέμα των PNR, των προσωπικών δεδομένων. Για μας την πολιτική μου ομάδα δηλαδή, είναι σαφές ότι θέλουμε αποτέλεσμα. Θέλουμε ασφάλεια των πολιτών μας που μετακινούνται ως επιβάτες ε, προς την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Θέλουμε λοιπόν την ασφάλειά τους. Θα πρέπει και εσείς όμως να κατανοήσετε και γι' αυτό σας παρακαλώ να το σκεφτείτε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε καθορίσει νέες θεμελιώδεις αξίες στην Ευρώπη και οι ημερογνώμονες, οι νομομαθείς μας, μας λένε ότι τα αποτελέσματα που είχαμε επιτύχει στι συζητήσει πριν από τις θερινές διακοπές δεν είναι επαρκή, δεν ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες που ε, υπαγορεύουν, που θεμελιώνουν οι νέες ε, διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε λοιπόν ακόμη απόσταση. Ζητώ λοιπόν την κατανόησή σας ότι και εμείς έχουμε τις αρχές μας, τις έχουμε καθορίσει στη συνθήκη της Λισαβόνας και οφείλουμε να τις σεβαστούμε. Μια δεύτερη σκέψη για το δεύτερο ντοσιέ που είναι ε, η, συνθήκη η συμφωνία μάλλον πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, θα δούμε και στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες δεκαετίες ότι χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο ανταλλαγή δεδομένων για τον αγώνα κατά της ε, ε, οργανωμένης εγκληματικότητας που λαμβάνει όλο και πιο διεθνείς μορφές συνεργασίας θα είναι μεγάλη ευκαιρία αν επιτύχουμε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή δεδομένων, αλλά πρωτίστως στον καθορισμό προτύπων για την ανταλλαγή αυτή δεδομένων διεθνώς, γιατί τότε μπορούμε χέρι με χέρι να προχωρήσουμε μαζί. Παρακαλώ να το δείτε και εσείς αυτό ως ευκαιρία. Το τελευταίο που είναι η λεγόμενη cyber security, θα ήθελα ε, να ρωτήσω πού βλέπετε, μάλλον πού θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει, σε, ποια, σε ποιο σημείο πρόοδου δηλαδή, θα χρειαστεί περισσότερη ε, συνεργασία και περισσότερη δέσμευση υπέρ μια συνεργασία και από τι δύο πλευρέ, οι ΗΠΑ και η Ενωμένη Ευρώπη. Η κυρία Λόπεθ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και η ομάδα μου επίσης ε, εκφράζει την αλληλεγγύη της και, συμφωνεί, και υποστηρίζει τον Αμερικανικό λαό για αυτό το τρομοκρατικό πλήγμα της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Και θέλουμε να αξιολογήσουμε και να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα οποία στην αμοιβαία δικαστική αρρωγή είναι θετικά. Όλα τα, όλες τις θετικές επιπτώσεις για την αμοιβαία συνεργασία μας. Ωστόσο από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο αληθεύει είναι ότι υπάρχουν μεταξύ άλλων διαφορετικές προσεγγίσεις και έννοιες για το τι είναι ιδιωτική ζωή και προσωπικά δεδομένα και διαφορετική επικέντρωση από αυτών των θεμάτων ιστορικά όσον αφορά την παράδοσή μας. Αυτό το οποίο είπε για το ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει έλλειψη προστασίας ε, δεδομένων, για μας τους Ευρωπαίους βουλευτές ε, και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους δεν συμβαίνει αυτό. Για μας η ιδιωτική ζωή, η ιδιωτική σφαίρα είναι ένα δικαίωμα χωρίς προϋποθέσεις και όρους επισκέφθηκα τις Ηνωμένε Πολιτείε και για τους Αμερικανούς η ιδιωτική ζωή, ιδιωτική σφαίρα είναι υπόρους και προϋποθέσεις δικαίωμα σε όλη την ομολογία και νομοθεσία τον είπα. Και γι' αυτό σε καταστάσεις όπως αυτές που έζησε ο Αμερικανικός λαός, αλλά και οι Ευρωπαίοι επίσης, υπήρξαν περιορισμοί εγγυήσεων. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας τώρα πρέπει να σέβεται το κράτος δικαίου και την ένωμη τάξη. Γι' αυτό υπό το δικό μας πρίσμα υπάρχει μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλυφθεί ακόμα. Και υπάρχουν ακόμα προβλήματα τα οποία πρέπει από κοινού να επιληθούν. Αληθεύει ότι είναι δύσκολο, δυσχερές αυτό το εγχείρημα, γιατί τα εγκλήματα της ε, εγκληματικότητας, ε, του οργανωμένου εγκλήματος κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, έχουν εδώ και ένα συλλογικό ε, ορισμό και έννοια, καθώς επίσης και διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τους ορισμούς, όσον αφορά τις νομολογίες και τις νομοθεσίες μας. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Γενικός Εισαγγελέας, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας των πολιτών μας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών μας, ακόμα και των δικονομικών εγγυήσεων όσον αφορά τους ε, υπόπτους ε, κάποιων, ε, συντέλεσης κάποιων πράξεων. Εδώ εξακολουθούν να υπάρχουν αποστάσεις ε, που μας χωρίζουν. Γιατί ακόμα οι αξίες μας έχουν πολύ μεγάλη απόσταση που τις χωρίζει από το πώς ε, αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πώς επικεντρωνόμαστε εμείς ως Ευρωπαίοι σε αυτά. Ενώ αποθηκεύονται και διατηρούνται στοιχεία επί τόσα πολλά χρονικά έτη. Ενώ υπάρχει η εκπόνηση των στοιχείων τρομοκρατών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο για να καταλήξουμε σε μια γενική συμφωνία επ' αυτών. Ευχαριστώ. Uh, θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον uh, Γενικό Εισαγγελέα στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι που είστε ανάμεσά μας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι συμμεριζόμεθα την αποφασιστικότητά σας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Χαίρομαι λοιπόν γιατί υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Eurojust και τη Europol. Είναι ευρωπαϊκές υπηρεσίε που εμείς δημιουργήσαμε και θα θέλαμε να τις βλέπουμε να δραστηριοποιούνται καλύτερα. Απ' την άλλη δεν εκπλήσει κανένα όταν βλέπει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία του ιδιωτικού χώρου γενικότερα. Δεν συμφωνώ μαζί σας για το ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην πραγματικότητα και όχι σε υποθέσεις, γιατί η ίδια η φιλοσοφία, αν θέλετε, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι να αποφύγουμε τα λάθη ή ιδιαίτερα τα λάθη ερμηνείας της ισχύουσας τοποθεσίας. Σε αυτή τη φάση λοιπόν είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί από ό,τι συνήθως, διότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι πλήρως από τη συμφωνία TFTP. Έχω, δεν θέλουμε εμείς την μεταφορά χίδιν δεδομένων, θέλουμε επιλεκτικές μεταφορές, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται μέχρι τώρα και ε, δεν εκπλήσωμε γιατί οι διαπραγματεύσεις για το PNR και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι διμερείς συμφωνίες δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα. Αυτό είναι κάτι που δεν με εκπλήσει. Ε, βέβαια σέβομαι το ότι εσείς θα θελήσετε να κάνετε αυτό το οποίο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο για τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Αμερικανό πολίτη. Από την άλλη εμείς θα πρέπει τα παράπονά μας εισαγωγικά να τα στρέψουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτοί εκπροσωπούν την Ευρώπη και είναι ο ομόλογός σας θα έλεγα σε αυτές τις επαφές. Δύο μικρές ερωτήσεις σχετικά με την εντολή που έχετε. Θα ήθελα θα το εκτιμούσα να μας πείτε αν επί τη βάση του πατριωτικού νόμου, του Patriot Act, οι Αμερικανικές αρχές έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία ε, είναι σωρευμένα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν όμως την έδρα τους στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεύτερη ερώτηση. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για κάποιες διατυπώσεις στις διμερείς συμφωνίες επαρκής κίνδυνος, εθνικός κίνδυνος. Ε, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Ποιες είναι οι νομικές εγγυήσεις και οι δυνατότητες αποκατάστασης ε, του δικαίου σε περίπτωση υπερβολών. Για τους πρασίνους ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ το Γενικό Εισαγγελέα. Σας ευχαριστώ που είστε ανάμεσά μας. λέει ο κύριος Άλμπρεχτ Χαίρομαι λοιπόν που είστε ανάμεσά μας. Ελπίζω να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τους ομολόγους μας στις Ηνωμένε Πολιτείε όταν πάμε πια εκεί και εσείς όταν ξαναέλθετε, ξαναέλθετε εδώ. Θέλουμε να συναντάμε όλο και περισσότερο τα μέλη του Κογκρέσου, ιδιαίτερα όταν μας επισκέπτονται εδώ στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή ή μάλλον βρισκόμαστε ακριβώς σε μια ιστορική καρδί εδώ και μια δεκαετή περίπου περίοδο. Έχουμε μοιραστεί κοινέ εμπειρίες με τις τρομοκρατικές επιλές και τις απειλές του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως είπατε, όπως ακούστηκε, σεβόμαστε τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε η στιγμή όμως παραμένει ιστορική γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας ακόμα περισσότερο. Πολλές από τις συμφωνίες τις οποίες συνήψαμε όλα αυτά τα χρόνια οφείλονται στους κοινού στόχους τους οποίους έχουμε και οι κοινοί αυτοί στόχοι συνεχίζουν να παραμένουν κοινοί. Αν και βέβαια έχουν αναφανεί κάποιες διαφορές στην διαπραγμάτευση θεμάτων όπως των εγγυήσεων για τον ιδιωτικό χώρο και σε αυτή τη φάση την ιστορική μπορούμε, έχω την αίσθηση, να φτάσουμε σε κοινά επίπεδα, μπορούμε να φτάσουμε σε κοινού κανόνες, γιατί όχι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους συμπολίτε μας. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει στους ευρωπαϊκούς λαούς ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγγυήσει σχετικά με την προστασία των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και με την ισορροπία των εξουσιών και την ισορροπία των σχέσεων κράτους-πολίτη. Όταν βλέπει κανείς το σφαιρικότερο περιβάλλον στο οποίο κινούμεθα σε αυτή τη φάση, διαπιστώνει ότι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις οι οποίες κυρίως είναι κοινέ προκλήσεις. Από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπε χώρες του κόσμου σέβονται αυτά τα οποία εμείς σεβόμεθα. Και γι' αυτό ακριβώς τα θεμέλια της συνεργασίας μας θα πρέπει να ενισχυθούν με την υιοθέτηση νέων μέτρων όπως ε, το κοινά πλαίσια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και σαν εισηγητής θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεργαστείτε ακόμα περισσότερο με μας και να θεωρήσετε ότι είναι μια εκκίνηση η συμφωνία αυτή για ένα νομοθετικό διατλαντικό πλαίσιο το οποίο δεν έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, αλλά παρόλα αυτά οι προκλήσεις παραμένουν οι ίδιες και είναι κοινέ. Λοιπόν, θα υπάρξει ένας πρώτος γύρος τώρα απαντήσεων από τον κύριο Χόλτερ. Και θα ετοιμαστούν έτσι τα υπόλοιπα μέλη που θα πάρουν το λόγο για ένα λεπτό ο καθένας, αλλά έχει το λόγο Γενικός Εισαγγελέας. Και εγώ προετοιμαστήκαμε για την έλευσή μας εδώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκφραση ε, συμπάθειας και κατανόησης την οποία εκφράσατε σχετικά με την 9η Σεπτεμβρίου. Ε, έχω σημειώσει κάποιες από τις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε. Η, εικόνα που έχουμε, η ιδέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες είναι διαφορετική από ό,τι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον μας, ε, είτε οι τρομοκράτες ε, είτε οι εγκληματίες, δεν σέβονται τα σύνορά μας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ε, ποια είναι τα θέματα τα οποία τίθενται εντός των σύνορων μας, να ορίσουμε κάποια τεχνικά προβλήματα και θέματα πέρα από τις κοινέ μας αξίες, οι οποίες παραμένουν όπως είπα κοινέ στην προκαταρτική μου παρατήρηση. Ε, σαφώς και ε, εμείς αξιολογούμε θετικά τα προσωπικά δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ε, τα προστατεύουμε με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους μηχανισμούς με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και γι' αυτό ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν απέχουν τόσο πολύ μία από την άλλη. Για τα PNR να πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μέχρι το Μάιο που καταλήξαμε σε μια συμφωνία, το συμφωνία ισχυρότερη από το κείμενο του 2007 όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το PNR, οι οποίες βέβαια ακόμα συνεχίζονται. Να υπογραμμίσω ότι είναι βασική μας επιθυμία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες όλες τις σωστές απαντήσεις. Εμείς ερχόμαστε εδώ ανοιχτοί και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας σε επίπεδο ισότιμων εταίρων. Θα υπάρξουν βέβαια διαφορές μεταξύ μας, θα υπάρξουν καλύτερες ιδέες από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι από τις Ηνωμένες Πολιτείες μερικές φορές, αλλά από την άλλη μπορεί να ισχύει και το αντίθετο ελπίδα μας είναι ότι μέσα από την διαπραγμάτευση, μέσα από την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε φίλους και ισχυρούς συμμάχους, σε ισχυρούς εταίρους θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αμοιβαία επωφελές και αμοιβαία συνεκτικό με τις βασικές μας αρχές και νομίζω ότι καμία βέβαια από τις δύο πλευρές δεν θα μείνει πλήρως ικανοποιημένη, απόλυτα ικανοποιημένη. Αλλά παρόλα αυτά όλοι θα έχουμε σαν στόχο να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από αυτούς οι οποίοι όπως είπα δεν σέβονται τα σύνορά μας, δεν σέβονται τις βασικές μας αξίες και δεν σέβονται τις επιθυμίες και την ψυχή των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ για την συγκεκριμένη και ξεκάθαρη απάντηση. Τώρα περνάμε στον δεύτερο γύρο θα ήθελα όμως να μην μιλάτε πάνω από ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί όπως σας είπα θα είμαι απόλυτος. Και ως Βος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα χρειαστεί να βάλετε τα ακουστικά. Και από τη δική μου πλευρά, λοιπόν, ευχαριστίες για την έλευσή σας εδώ Μα ενδιαφέρει πολύ η ανταλλαγή απόψεων, ώστε να παραμείνουμε στη συζήτηση. Πολλά από τα ερωτήματα μου ήδη καλύφθηκαν. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστώ σε δύο μόνο συγκεκριμένα ε, θέματα. Αφενός και βεβαίως ο κύριος Πρέσβης και οι συνεργάτες του ε, εργάζονται πολύ καλά επ' αυτού. Θα προχωρούσαμε νομίζω στο PNR εάν ρίξουμε ιδιαίτερα το βάρος μας στο πεδίο εφαρμογής όσο και αν είναι δυσχερείς οι λεπτομέρειες λόγω των εσωτερικών κατανομών της ε, δικαιοδοτικής αρμοδιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι βέβαιος ότι οι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν την επινοητικότητα να δώσουν τις λύσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο, θα ευχαριστήσω βεβαίως πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις υποδείξεις που έγιναν για τις συλλήψεις και οδήγησαν μάλλον στις συλλήψεις στο Βερολίνο σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων αλλά και τη ρύθμιση του διαδικτύου, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε κοινά πρότυπα. Αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο και εντονότερα. Ευχαριστώ. Κράισλερ Ντόφλερ των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το 2006-2007 λειτουργήσε μια έκτακτη επιτροπή η οποία είχε συζητήσει τότε τις ε, έκτακτες εκδόσεις το, τις extraordinary renditions των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θέλω να μάθω τα δεδομένα αυτά σε ποιους πήγαν, διότι είχαν γίνει τότε απαγωγές με ε, λάθος, ε, λάθος, σε βάρος λάθος προσώπων. Αλμάσρι στη Γερμανία, Μαχέρ Αρά από τον Καναδά. Πώς μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι με τα δεδομένα PNR και όλα τα άλλα δεδομένα που συλλέγεται δεν θα επαναληφθούν γεγονότα όπως εκείνα που έγιναν, που σημειώθηκαν τότε επί Προεδρίας Bush. Έρχεται για παράδειγμα η Πακιστανική Υπηρεσία Πληροφοριών και σας προσφέρει δεδομένα ή η Ισραηλή Μοσάντ. Έχω μεγάλες επιφυλάξεις σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων αυτών. Και βρισκόμαστε στο πεδίο εντάσσεως ανάμεσα στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να προστατεύσουμε την προσωπική σφαίρα και τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Λάθη θα γίνονται, αλλά τέτοιου είδους λαθροχειρίες δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Πράσινη, Ταβάρες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε ε, Υπουργέ. Αναφέρατε ορισμένες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, της Μαδρίτης και επίσης της Αμπούζα. Περίμενα να ακούσω και για το Όσλο στην Νορβηγία. Παρόλο που είναι πολύ διαφορετικές οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις, θα πρέπει, τη θυμηθήκαμε εμείς, συζητήσαμε στην Ολομέλεια και οι περισσότερες από τις πολιτικές μας ομάδες θεωρούν ότι αποτελούν και ε, την κατάληξη μιας δεκαετίας Ισλαμοφοβίας και μιας ε, μεγάλης επιθετικότητα απέναντι στον αλλοδαπό, τον ξένο. Πρέπει βέβαια να αντιμετωπίσουμε τις ε, επιθέσεις αυτές με διαφάνεια, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις λησμονούμε. Τώρα, πρακτικά ερωτήματα. Δεν είναι παράνομο να παρακολουθούνται τα τηλέφωνα ξένων αλλοδαπών πολιτών στις ΗΠΑ. Δεύτερο, εσείς ως μέλος εκτελεστικής εξουσίας θεωρείτε ότι το Privacy Act πρέπει να επεκταθεί και στους ξένους πολίτες. Τρίτο, μπορούν να διατηρηθούν οι συνταγματικές διατάξεις χωρών όπως της δικής μου, ώστε να μην δίδονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες όπου μπορεί να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Σε πρόσφατη ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας ακούστηκε ότι εταιρείε με έδρα και στην ΗΠΑ και στην Ευρω... Ε, Ευρώπη μπορεί να έχουν ίσως ε, συγκρουόμενες υποχρεώσεις ε, αποκάλυψη ή μη δεδομένων. Εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση συγκρούσεως, ποια υποχρέωση θα πρέπει να έχει προτεραιότητα, υπεροχή αυτή απέναντι στις ΗΠΑ ή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω επίσης ότι το Ομοσπονδιακό Δίκαιο στις ΗΠΑ προστατεύει την προσωπική σφαίρα των Αμερικανών πολιτών, όχι όμως μη Αμερικανών πολιτών, για παράδειγμα Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης, παρόλο που η προσωπική σφαίρα προστατεύεται μέσα στα πλαίσια τη Συμφωνία Ευρώπη, Αυτέ οι συμφωνίε δεν έχουν την ισχύ νόμου και γι' αυτό δεν είναι εκτελεστέ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χόλτερ για την παρουσία του. Είχα τη δυνατότητα να τον συναντήσω στη Washington στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων Σύντομα τώρα, μιλήσαμε για πολλές αντιθέσεις στον τρόπο που καταπολέμησε τη τρομοκρατίας. Τις τελευταίες μέρες έρχεται στην, στο φως η πρώτη έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα και για την ομογενοποίηση των νομικών βάσεων των τρόπων αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέματα ανείχνευσης ή ανιχνευσιμότητας των χρηματοδοτικών μέσων, ε, εξέταση γενικά όλων των διοικητικών στενών σχέσεων ανάμεσα σε εγκληματικά στοιχεία κτλ. Τι πιστεύετε εσείς στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος μπορούμε να κάνουμε από κοινού στι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας είπε ένα λεπτό από σοσιαλιστές. Κύριε Γενικέ Εισαγγελέα. Θα σας πω ότι ε, όταν ήμουν πολύ νέος γνώρισα τον Ρόμπερτ Κέννεντι που ήταν εκείνος ο οποίος είχε το αξίωμά σας πριν από πολλά χρόνια και ως ακόλουθος της ε, αμερικανικής πολιτικής αναφέρατε τον πρόεδρο Ομπάμα σε σχέση με το βαθμό στον οποίο καταφέρνετε να ε, δώσετε ε, μία διάσταση στον αγώνα αυτό ε, που ακολουθείτε για τους Ευρωπαίους. Το πνεύμα όμως του Ομπάμα είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο ίσχυε στο παρελθόν. Και επίσης όσον αφορά τους βουλευτές και στο Κογκρέσο και στον κοινοβουλευτικό κόσμο θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη διαφορά αυτή και τις επιπτώσεις που έχει στον κοινοβουλευτικό κόσμο. Ε, Προσέξτε, πριν από λίγες μέρες ε, θυμηθήκαμε τα θύματα της 11 Σεπτεμβρίου 2001 και με όλους αυτούς ε, εκείνους που έχασαν τη ζωή τους υπέρ της ελευθερίας. Αυτά τα θέματα συζητάμε. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Όμως με την ταπεινή μου γνώμη ως θύμα τρομοκρατία, θα έπρεπε να σα πω το πιο σημαντικό, το πιο το ανώτατο δικαίωμα που έχουμε ενώπιον μας είναι το δικαίωμα στη ζωή και θα πρέπει να ενδιαφερθούμε να προστατέψουμε τη ζωή των πολιτών μας. Η κύρια, το κύριο μέλημα της ομάδας μας είναι το εξή. Σε σχέση με τις συναντήσεις με τους Αμερικανούς είχαμε τα παράπονα να εξευρεθεί ένας εταίρος αναφέρθηκε με αποτελεσματικό τρόπο είπαν οι Αμερικανοί για τους Ευρωπαίους. Όταν ήθελαν να έρθουν σε επαφή με τους Ευρωπαίους δεν γνώριζαν με ποιον έπρεπε να έρθουν σε επαφή και ε, πώς να τον καλέσουν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι γίνεται σε σχέση με την προστασία ακριβώς των θυμάτων της τρομοκρατίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η κυρία Μπορσελίνο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, δόκτωρα Όλτερ, που είσαστε μαζί μας. Αναφερθήκατε σωστά στην τρομοκρατία, αναφερθήκατε και στο οργανωμένο έγκλημα, δεν αναφερθήκατε στη μαφία. Μαφία είναι ένα ιδιαίτερο θα έλεγα σχήμα εγκληματική δραστηριότητας και γνωρίζεται στι ΗΠΑ περί τίνο πρόκειται. Τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, η συνεργασία με το Υπουργείο δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ιταλική δικαιοσύνη, τους Ιταλούς δικαστές ε, Μπορσελίνο, Φαλκόνε, ήταν ιδιαίτερα καλές ε, οι σχέσεις ε, και ιδιαίτερα καρποφόρες. Υπάρχει σε αυτή τη φάση συνεργασία. Είναι χρήσιμη. Και ε, τι χώρος θα έλεγα δίδεται στην καταπολέμηση μιας διεθνικής πολλαπλής εγκληματικής δραστηριότητας όπως η μαφία. Τον λόγο τώρα κύριε Γενική Αγγελέα. Επιτρέψτε μου να πω ότι η αμφίδρομη δράση με τα μέλη της ε, ομάδας δεν είναι ανώμια με εκείνη της επαφής ε, με τα μέλη του Κογκρέσου στη ΣΥΠΑ Διαφορετικά οι ερωτήσεις σας πρέπει να πω ήταν πιο στοχοθετημένες και ένα το πω νέο σκηνικό για μένα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα εδώ που έχουμε μπροστά μας. Για κάποια από αυτά ο α, πρέσβης α, τον είπα στο Βέλιο θα ε, στις, ευρωπαϊκές κοινότητες θα τοποθετηθεί. Για τις ε, συλλήψεις και εκδόσεις ε, rendition για το 2006 που ε, τον καιρό εκείνο είτε είχε διαφορετική ε, θέση, για παράδειγμα ε, είχαν διαφορετική θέση οι ΕΠΑ όσον αφορά την κυβέρνηση Μπούς για παράδειγμα και την κυβέρνηση Ομπάμα. Έχουμε μια διαφορά όσον αφορά την συνέχεια της παράδοσης με την προηγούμενη κυβέρνηση και είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό το πλαίσιο και είπαμε και αναφέραμε ότι μπορεί να έκαναν σφάλματα οι ΕΠΑ στο παρελθόν ή να φέρθηκαν με έναν τρόπο που δεν συνείδε με τις αρχές εκείνες τις οποίες θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Προσπαθήσαμε την κυβέρνηση Ομπάμα να κλείσουμε ε, το Γουαντάναμο και για την κατάργηση κάποιων τεχνικών, ιδιαίτερα όσον αφορά για παράδειγμα τα βασανιστήρια και τα οποία δεν θα έπρεπε να συνεχιστούν και υπήρξε μια διαφορά, μια καμπή ας το πω έτσι, σε σχέση με εκείνα τα οποία συνέβαιναν στο παρελθόν και που ήταν για παράδειγμα απαράδεκτα και δεν μπορούσαν να συνεχιστούν υπό την κυβέρνηση Ομπάμα, υπό τον πρόεδρο Ομπάμα. Τώρα για το Όσλο, αυτό το οποίο συνέβη εκεί αν είναι αποτέλεσμα Ισλαμοφοβίας ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε σε αυτή τη μάχη κατά της τρομοκρατίας που δίνουμε. Ότι για παράδειγμα εμείς στη ΣΥΠΑ και από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, προσπαθήσαμε να έχουμε επαφή με τους ε, ε, μουσουλμάνους ε, στις ΗΠΑ ε, για να δείξουμε ότι τους σεβόμαστε και ότι τους ξεχωρίζουμε σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν είναι αυτή ο στόχος μας. Η τρομοκρατία συνδέεται δεν είναι κάτι το οποίο να συνδέεται με συγκεκριμένη θρησκεία. Το Ισλάμ είναι μια πολύ μεγάλη θρησκεία. Υπάρχουν όμως κάποιοι που χρησιμοποιούν αυτή τη θρησκεία για να εξυπηρετήσουν ιδιωτελώς κάποιους ε, σκοπούς και στόχους δικούς τους. Και έτσι βλέπουμε ότι γίνεται κατάχρηση της ε, θρησκείας αυτής. Ε. Και αυτό που βλέπουμε τώρα πρέπει υπό αυτό το πνεύμα να εξεταστεί. Όσον αφορά τώρα την... Να κοιτάξω μια στιγμή τις σημειώσεις μου. Την θανατική ποινή αναφέρθηκε και τα προσωπικά δεδομένα. Στη ΣΥΠΑ όταν έχουμε θέμα έκδοσης ε, ατόμων από μια άλλη χώρα που δεν έχει τη θανατική ποινή ή σε σχέση με το θέμα της θανατικής ποινής ε, μέσα στο πλαίσιο των είπα συχνά ή θα έλεγα κιόλας γενικά θα λέγαμε αν το θέτει αυτό το θέμα μια χώρα για την έκδοση αυτού του ατόμου στη ΣΥΠΑ, αυτό δεν θα αποτελέσει, ας το πω έτσι, αντικείμενο της ε, ε θανατικής ποινής. Θα σεβόμαστε αρχές ε, κατανοούμε ότι υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ ΙΠΑ και πολλών χωρών όσον αφορά αυτές τις ε, πτυχές για το θέμα της θανάτικης ποινής. Για να δω μια στιγμή στη συνέχεια. Uh, Κάνουμε λόγο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, οργανωμένης εγκληματικότητας. Και πριν από κάποιες εβδομάδες σε σχέση με την συνάντηση που είχαμε, με την κυβέρνησή μας ότι η τρομοκρατία αναλώνει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειές μας. Δεν έχουμε όμως ε, αγνοήσει, δεν αμελούμε το γεγονός ότι ε, το οργανωμένο έγκλημα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και είναι κιόλας και προτεραιότητα για τι ε, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Καλωσορίζω και χαιρετίζω τις παρατηρήσεις που έγιναν όσον αφορά το πνεύμα του Προέδρου Ομπάμα και το πνεύμα στο παρελθόν του Ρόμπερτ Κένεντι ως Υπουργού Δικαιοσύνης, ως Attorney General Γενικού Εισαγγελέα στις ΗΠΑ. Ήταν υπόδειγμα, είναι ο προσωπικός μου ήρωας. Έχω πολλές φωτογραφίες ε, δικές του στο γραφείο μου και έχω την ελπίδα ότι διεξάγουμε τις εργασίες μας υπό το πνεύμα και την έννοια με την οποία εκείνος ε, δρούσε και προσέγγιζε αυτά τα θέματα. Και ελπίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα φέρεται και συμπεριφέρεται με τρόπο που προσεγγίζει και είναι παρόμοιος με τον αδερφό του Ρόμπερτ Κέννεντι, τον Τζον Κέννεντι, τον πρόεδρος τον είπα πριν από τον Ομπάμα. Και έχουμε εδώ και τα θέματα ασφάλειας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια ένταση, ένα πεδίο έντασης μεταξύ των αρχών και αξιών μας, αυτά που θέλουμε να προστατεύσουμε όσον αφορά την ελευθερία και την προστασία των πολιτών μας και την έννοια της ασφάλειας που θέλουμε να προστατεύσουμε από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει αντίφαση. Υπάρχουν τρόποι να προστατεύσουμε τους πολίτες μας παραμένοντας πιστοί στο σεβασμό των αρχών και αξιών μας χωρίς να απεμπολούμε αυτές τις αξίες και σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ υπήρχαν διαφορές. Δεν έχουμε εμεί αυτές τις απόψεις όπως η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έχουμε την άποψη ως πρόεδρος Ομπάμα ή ως υπουργό Δικαιοσύνης. Μπορούμε να σεβόμαστε τις αρχές των δικαιωμάτων των πολιτών μας και των Ευρωπαίων πολιτών όπως ε, είναι σεβαστές αυτές οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως να προστατεύουμε την ασφάλειά τους. Και για την εφαρμογή όσον αφορά διατάξεις ε, της Συμφωνίας PNR ε, προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτών θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πρέσβη. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ. Απλά πολύ σύντομα. Κύριε Φως, ρωτήσατε τι συμβαίνει με τα PNR και τη συμφωνία αυτή. Όπως ανέφερε πιο πριν από ό,τι άκουσα ο Γενικός Εισαγγελέας, από πλευρά Jane Honglu, ε, υπεύθυνων διαπραγματεύσεων και από την, ε, ε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης που θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα για αυτά τα θέματα. Πολλή δουλειά έχει γίνει ήδη. Καθίσαμε στο διαπραγματευτικό τραπέζι επί μεγάλο χρονικό διάστημα και από πέρυσι μέχρι σήμερα. Οι συζητήσεις εξελίσσονται και συνεχίζονται βέβαια. Δεν έχουμε φτάσει στην λειτουργική φάση εφαρμογής ακόμα. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω και εσάς κύριε Φως και τα άλλα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κάνατε σκληρή δουλειά. Ήρθατε στη Washington αρκετοί από εσά για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία αυτής της ε, Passenger ε, Name records συμφωνίας και να δείτε πώς θα λειτουργούν τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προσπάθειες και σας ευχαριστούμε για αυτές. Απομένει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον συνάδελφο και που ο κύριος Μπρουσ Σουόρτς θα μπορέσει να αναφερθεί σε αυτά πιο εξειδικευμένα. Σας ευχαριστώ πρέσβη και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ευκαιρία που δίνετε. Από πλευρά τον είπα σε αυτή την συμφωνία φυσικά εξετάσαμε στις συζητήσεις μας αρκετά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα. Θα ήθελα σύντομα πρώτα να αναφερθώ στο νομοθέτημα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αναγνωρίζουμε ότι σε σχέση με αυτό το θέμα δημιουργούνται κάποια θέματα. Όμως να τονίσω ότι όπως ακούσατε και προηγούμενα, στο πρακτικό επίπεδο εφαρμογής δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ πολιτών ΗΠΑ και πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ιδιωτική ζωή και τις διατάξεις για την, ε, το σεβασμό και εφαρμογή του νόμου. Ακόμα και για θέματα δικαιοσύνης ε, που ε, αντιμετωπίζουν ένα ειδικό πλαίσιο. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχουν διαφορές, δεν υπάρχει αρνητική διακριτική μεταχείριση όσον αφορά υπηκός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά η κάλυψη η νομική διασφαλίζεται ώστε να δούμε ποιου είδους στοιχεία έχουν αποθηκευτεί και να δούμε ποιες ε, εξαιρέσεις ε, από πλευράς της ε, Freedom Act υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως αρνητική μεταχείριση εις βάρος πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για την πρόσβαση όσον αφορά τους παρόχους στο διαδίκτυο και τα ε, αρχεία που κρατούνται. Δεν υπάρχει διαφορά για την προσέγγιση που υιοθετείται από τη ΣΥΠΑ και από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε πολλά για την Patriot Act, αλλά αυτά είναι παραπλανητικά όσον αφορά την εφαρμογή. Πράγματι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την θέση ότι έχει δικαίωμα να έχει τα στοιχεία εκείνα των θηγατρικών εταιριών που βρίσκονται στη δική της επικράτεια στη διάθεσή της. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είπαμε, μέσα στο Patriot Act, ότι οι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο να ε, έχουν ε, δυνατότητα άντλησης αυτών των ε, στοιχείων. Έχουμε όμως ε, την ε, διαφοροποίηση και για έναν πάροχο υπηρεσιών στο διαδίκτυο όταν ε, μπορεί να γίνει, να διατυπωθεί το αίτημα σε έναν τέτοιο πάροχο να δώσει στοιχεία για στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί και κρατούνται στη ΣΥΠΑ. Βλέπουμε εδώ σε σχέση με τους υπηκόους ε, των κρατών ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των υπηκών ΙΠΑ ε, ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Και το άλλο το οποίο ήθελα να πω είναι το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων το οποίο ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας πιο πριν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους πολίτες τους μπορεί να, σε τέτοιου είδους παρακολουθήσεις να ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. Εμείς λέμε ως είπα ότι δεν είμαστε τέλειοι Απλά λέμε ότι κάθε ένα από τα συστήματά μας στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύει την ιδιωτική ζωή και σφαίρα με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι το ουσιώδες παρά τις διαφορές ή αποκλήσεις μας. Σας ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσει θα λάβει τον λόγο ο Γενικός Εισαγγελέας. Ένα που πρόσεξα στις σημειώσεις μου είναι το θέμα της αποζημίωσης για τα θύματα ως παρατήρηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό στη ΣΥΠΑ τα τελευταία χρόνια. Πάντα πρέπει να λογοδοτούν και να είναι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα που έχουν ε, ε, διαπράξει ε, άτομα. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε επίσης και τα θύματα και να δούμε ένα ολόκληρο φάσμα δυνατοτήτων που θα στοχεύουν και θα σχεδιάζουν όχι μόνο την οικονομική συνιστόσα αυτών που έχουν υποστεί τα θύματα, αλλά συνολικά να δούμε την ζημιά που έχουν υποστεί έτσι με συγκεκριμένους μηχανισμούς που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα άτομα που ήταν αντικείμενο ως θύματα της τρομοκρατικής πράξης ε, της 11 ε, ε, Σεπτεμβρίου 2001 εν μια ολόκληρη αλυσίδα μέτρων αυτό αντανακλά ακριβώ από πλευρά των ΙΠΑ την προσπάθεια να γίνει κατανοητό ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην εφαρμογή και σεβασμό του δικαίου και των διατάξεών του, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε μόνο τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες, πρέπει να προστατεύουμε και να λαμβάνουμε υπόψη εκείνους που υπήρξαν και ήταν θύματα αυτών των τρομοκρατικών πράξεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Εισαγγελέα. Ευχαριστούμε. Το συμπέρασμα τέλος τέλος αυτής της συζήτησης είναι προφανές θα έλεγα. Όλοι γνωρίζουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι διαφέρουν τα νομικά μας συστήματα. Το είδαμε μέχρι σήμερα σε αρκετές συζητήσεις. Αλλά είναι εξίσου προφανές ότι συμμεριζόμαστε την αποφασιστικότητα για την καταπολέμηση οποιοδήποτε εγκλήματος και τρομοκρατίας. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας το στένος να προστατευτούν τα θύματα οποιονδήποτε τρομοκρατικών πράξεων στην Αμερική, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στην Ουτόγια, οπουδήποτε και οποιασδήποτε μορφής. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές και πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές των νομικών μας συστημάτων για να πετύχουμε κοινούς στόχους που έχουμε ενώπιον μας. Σας ευχαριστώ για αυτή την έκφραση καλών προθέσεων και σθένους και αποφασιστικότητας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Τελευταία αναγγελία. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το έργο μας το οποίο απομένει να καλυφθεί στην επόμενη εβδομάδα του Στρασβουργού στην περίοδο συνόδου στην Ολομέλεια και για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτές ε, τις ε, σημαντικές τοποθετήσεις ε, στον διατλαντικό ε, διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ θα υπάρξει μια συνάντηση των επαϊόντων που θα ε, συνέρθει στις 27 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες για να δώσουμε συνέχεια σε αυτά τα κεφάλαια όσον αφορά την εφαρμογή κοινέ ε, ερευνητικέ ομάδε ε, και θέματα ε, νομική και δικαστικής αρρωγή. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Εισαγγελέα που προσήλθατε. Είμαστε ευγνώμονε. Ευχαριστούμε.